E καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλημέρα σε διάφορες γλώσσες. Παρακαλώ, καθίστε. Περιμέναμε να γίνουν κάποιες τελικές διευθετήσεις για τις επικείμενες ψηφοφορίες. και φαίνεται ότι εντάξει και ο εξοπλισμός λειτουργεί, και παρακαλώ ησυχία. Έχουμε κάποιες ψηφοφορίες. Λοιπόν, αλλά να κάνω μια ανακοίνωση. κυρία Μακοβέ αποσύρει τις τροπολογίες 90 ε, και 93 που είχε υποβάλει. Βεβαίως έχουμε τώρα κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής ε, ΛΥΜΠΕ με την ε, ΚΟΝΤ. Είμαστε στην τελική φάση εξέταση, εξέτασης θεμάτων της αρμοδιότητάς μας. Και παρακαλώ ησυχία για να μπορέσουμε να συγκεντρωθούμε. Κύριε Πίρκελ, παρακαλώ. Κύριε Μέλλο, θα περιμένουμε. Λοιπόν, έχουμε κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής ε, Δημοσίων Ελευθεριών και ελέγχου του προπολογισμού με βάση το άρθρο 51 θα ψηφίσουμε για την καταπολέμηση των απατών ε, κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης μέσω ε, ποινικού νόμου. Η συγκίτρια είναι η κυρία Γκρέσλε από πλευρά τη Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού και εγώ από πλευρά τη Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών. Είναι συνέχιση της συνεδρίασής μας στις 20 Φεβρουαρίου. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία, εκτός αν οι εισηγητές δεν θέλουν να πάρουν το λόγο. Όχι, ωραία. Περνάμε λοιπόν απευθείας στην ψηφοφορία. Τροπολογία 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 και 51 ταυτόσιμες. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 και 49-50 από κοινού παρακαλώ κύριε Μέλλο. θέλετε ε, προφορική τροπολογία να υποβάλλετε Ναι, θα θέλαμε να υποβάλουμε μια προφορική τροπολογία. Να τη διαβάσω. Είναι η εξή. Το εισόδημα που προκύπτει από το ΦΠΑ θα συμπεριληφθεί στο πεδίο εφαρμογή τη οδηγία μόνο όσον αφορά τις περιπτώσει απάτης που έχουν διαμεθοριακή διάσταση. Πρόεδρος, υπάρχουν αντιρρήσεις για αυτή την προφορική τροπολογία. Α, υπάρχει αντίρρηση. Άρα δεν γίνεται δεκτή. Λυπάμαι κύριε μέλο. Υπήρξαν αντιρρήσεις από τέσσερα μέλη. Άρα σύμφωνα με τους κανόνες δεν γίνεται δεκτή. Ψηφίζουμε λοιπόν από κοινού τις 47, 49 και 50 όπως έχει συμφωνηθεί υπέρ παρακαλώ. Κατά ασαφές ε, να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. 15 υπέρ 32 κατά ήταν αρκετά σαφές. Απορρίπτεται. 52 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Αλλά ας ελέγξουμε. Ας ελέγξουμε. Ελέγχουμε λοιπόν. Πέρας. Ε, σαφώς, σαφώς. 53, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 4, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 με την προφορική τροπολογία. Υπάρχουν αντιρρήσεις για την προφορική τροπολογία. Όχι. Ωραία. Ψηφίζουμε. 54 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, οι υπόλοιπε καταπίπτουν και περνάμε στην 62 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 7 και 8 μαζί. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 9, 10 και 11 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 όχι καταπίπτει η 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται από ό,τι μπορώ να δω, αλλά ας ελέγξουμε. Έλεγχος ηλεκτρονικός. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. 23 υπέρ 24 κατά. Απορρίπτεται. 68 έως 71 υπέρ. Ε, από κοινού υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Ας ελέγξουμε γιατί ίσως είναι αμφίροπο. Άρχεται. Πέρας. Α, ανατροπή τώρα. 24 υπέρ, 23 κατά εγκρίνεται. 73 έως 76 από κοινού υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 77 υπέρ. Α, όχι, καταπίπτει. 78 και 79 από κοινού υπέρ. Κατά. Αποχές. Ασαφές, ας ελέγξουμε. Πέρας. 25 υπέρ, 23 κατά εγκρίνονται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Άσαφες. Έλεγχος. Βλέπω ότι υπάρχει διχογνωμία και ε, μεταξύ των ομάδων. Πέρα στις ψηφοφορίες. Δεκαεννιά με 29 απορρίπτεται. 82 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 84 υπέρ. Α, όχι. Α, όχι. Α, όχι, όχι. Ψηφίζουμε τον 84 υπέρ. Κατά Α, η 19 εγκρίθηκε. Α, από το 84 δεν μπαίνει στη ψηφοφορία. Και η 85. Α, όχι για το 85. Υπάρχει το δεύτερο τμήμα. Ωραία. Το δεύτερο τμήμα της 85 παρακαλώ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 86, 87 και 88 από κοινού υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται περνάμε στην 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Α, θέλετε να ελέγξουμε να ελέγξουμε λοιπόν την 91. Άρχεται ο έλεγχος. Πέρας. 30-19 εγκρίνεται. Περνάμε στην 94 υπέρ. Η 90 είπαμε έχει αποσυρθεί. 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 93 έχει αποσυρθεί 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 έχει ζητηθεί κατά τμήματα ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 Επίσης ε, ε, κατά τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 95 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Ω, είναι δύο, είναι δύο λατινικό. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Οπότε περνάμε στις ιδεολογικές ε, αναφορές, οι τροπολογίες 24, 25, 26, 29 και ένα ζουρί από κοινού, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εντάξει, ας ελέγξουμε. Ελέγχουμε αυτές τις πέντε τροπολογίες από κοινού. Υπάρχουν προβλήματα. Α, όχι, πέρα στις ψηφοφορίες. 27 με 23. Δεν Οι 27, οι 28 και 30 έχουν αποσυρθεί. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ζούρι 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 και 36 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 37 και 38 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ζουρί 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ζουρί 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 40 με την προφορική τροπολόγηση υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ζουρί 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α, όχι, απορρίπτεται, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ζούρι 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συγγνώμη, εγκρίνεται. Εγκρίνεται η 1. 43 με προφορική τροπολόγηση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα τελική ψηφοφορία ε, επί της τροποποιηθής εκθέσεως ονομαστική ωραία ψηφίζουμε άρχι. πέρασε 44 υπέρ, 2 κατά, 5 αποχές. Ευχαριστούμε τους εισηγητές. Ευχαριστούμε κυρία Γκρέσλα. Thank you. be the end of the joint meeting. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώθηκε η κοινή συνεδρίαση. The budget control. Ευχαριστούμε πολύ τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού που συμμετείχαν σε αυτήν την ψηφοφορία. Τώρα εμείς θα συνεχίσουμε με τη δική μας ε, ημερήσια διάταξη.